Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Βάσει της ημερήσιας διάταξης, η ψηφοφορία γίνεται βάσει της απροσταγμένης διαδικασίας για την έκθεση της κυρίας Σαρτόρη εν σχέση με την παράταση της συμφωνίας για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας. Ε, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη έκθεση της κυρίας Σαρτόρη εν σχέση με τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αλγερίας σχετικά με την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Εξάγεται ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στην Παρακαλώ. Λίνε. κύριος Λέινε έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμε κυρίε και κύριοι, θα ήθελα εξ ονόματο τη πολιτική μου ομάδα να ζητήσουμε για την επόμενη ψηφοφορία για την έκθεση Hefner να διεξαχθεί ω ονομαστική ψηφοφορία γιατί ήμουν στην ομάδα διαπραγμάτευσης και θα ήθελα να ξέρω πώς θα ψηφίσει ο καθένας. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποια αντίρρηση εν σχέση με την πρόταση αυτή που μόλις υποβλήθηκε. Εάν όχι, τότε θα προχωρήσουμε με ονομαστική ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στην ψηφοφορία τη έκθεση Hefner εν σχέση με τη διαβίβαση προ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον χειρισμό από αυτό διαβαθμισμένων πληροφοριών του Συμβουλίου πλην εκείνων του τομέα τη κοινή εξωτερική πολιτική και τη πολιτική ασφάλεια. Υπέρ παρακαλώ. Ονομαστική ψηφοφορία. Die Abstimmung ist geschlossen. Εγκρίνεται. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση Καρίμ. Πρόκειται για την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας και την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Λοιπόν, υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στην έκθεση Καντέκ. Συγγνώμη, παρακαλώ. Ποιο είναι το πρόβλημα. Κύριε ε, Πρόεδρε, είμαι συγγητής και θέλω να πω δύο λόγια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, μην ανησυχείτε, δεν πρέπει να χάσετε τα τρένα και τα αεροπλάνα σας. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε την ε, έκθεσή μου για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Ατλαντικό. Κοινοποιούνται σημαντικά μέσα για την ενδυνάμωση των εδαφών γύρω από τον Ατλαντικό. Υπάρχει και ένα οδικό χάρτη για την ε, βιομηχανική πολιτική για να ενισχύσουμε του στρατηγικού τομεί τη περιοχή του Ατλαντικού. Θα βοηθήσουμε έτσι και τι τον κλάδο της αλίας να αντιμετωπίσει την πρόκληση της παγκοσμιοποίησης. Χάρη σε εσά έχουμε δημιουργήσει ένα πραγματικό σχέδιο ε, ΜΑΡΣΑΡ για τον Ατλαντικό. Χρειαζόμαστε μια πραγματική πολιτική στην Ευρώπη για να ετοιμάσουμε την αυριανή ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε τον κύριο εισηγητή και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία της εν λόγω έκθεσης για την στρατηγική πολιτική συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή του Ατλαντικού. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά. Γίνεται δεκτή η έκθεση. Τώρα θα περάσουμε στην έκθεση του κυρίου David Martin για την εξαίρεση ορισμένων χωρών από τις εμπορικές προτιμήσεις. Έχουν κατατεθεί κάποιες ε, τροπολογίες. Θα ξεκινήσουμε με τροπολογία υπαριθμών 5 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στην Τροπολογία της Επιτροπής 1 ως 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία 6 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Η Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 της Επιτροπής. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Γίνεται δεκτή. Θα περάσουμε στην ε, τροποποιηθήσα, στο ψήφισμα υπέρ παρακαλώ, κατά αποχές θα πρέπει να γίνει επαλήθευση. Geschlossen. Πέρας της ψηφοφορίας ε, γίνεται δεκτό. Τώρα θα έρθουμε στο νομοθετικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Καρίμ για την ε, συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών στον ενεργειακό τομέα. Ξεκινάμε με την τροπολογία υπαριθμών 1 της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 4 των Σοσιαλδημοκρατών. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία ένα γάμα β της Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαλήθευση, εφόσον επιθυμείτε. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στο άρθρο 4, την τροπολογία της Επιτροπής, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και έτσι καταπίπτει την τροπολογία υπαρθμών 5. Και τώρα θα περάσουμε στο άρθρο 9, τροπολογία της Επιτροπής, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 2 καταπίπτει. Τροπολογία υπαριθμών 3. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Απορρίπτεται. Η τροπολογία της Επιτροπής υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Θα έρθουμε στο ψήφισμα έτσι όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα θα έρθουμε στην νομοθετική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια κύριε Καρίνς. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Γκαρθία Πέρες για συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα γεωργικά προϊόντα. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Απλώς ε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι σε σχέση με την τροπολογία παρθμών 103 παρουσίασαν οι πράσινοι πέρα από το ότι συμφωνώ πλήρω με το περιεχόμενο, ζητώ από την Ολομέλεια να την καταψηφίσει γιατί ξεπερνά τα όρια της συμφωνίας που, που πετύχαμε με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση. Αρχίζει λοιπόν η ψηφοφορία και θα έρθουμε στην απολογία υπερφών 104. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτει το μπλοκ 2 και θα έρθουμε στην τραπολογία υπαρθμών 103 που αναφέρθηκε με ονομαστική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία της ούτως τροποποιηθής πρότασης. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, νομοθετική ψηφοφορία, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία, πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Θερμά συγχαρητήρια κυρία Συγκήτρια. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Σοκόνη για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Έχουν ε, κατευθεί δύο τροπολογίες, η υπαριθμον δύο, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτει η δεύτερη τροπολογία της Επιτροπής και θα περάσουμε στην ψηφοφορία στην πρόταση έτσι όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία του νομοθετικού ψηφίσματος με ονομαστική ψηφοφορία. Ο εισηγητής ε, θέλει να πάρει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με βάλει το άρθρο 57 ζητώ η τελική ψηφοφορία του ψηφίσματος, του νομοθετικού ψηφίσματος, να μην γίνει σήμερα. Θα ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα ψηφίσουμε και αυτή την πρόταση της ίδιας. Ποιος είναι υπέρ της αναβολής. Κατά. Αποχές. Η πρόταση γίνεται δεκτή. Παρακαλώ κύριε Λάμπερτ. Θα περάσουμε στη δική σα έκθεση. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είμαστε στην ίδια κατάσταση, η Σοφή και εγώ, και για αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ την προσοχή στο ότι είναι μια έκτακτη περίπτωση αυτή. Μετά από μια επιτυχή ολοκλήρωση του τριμερούς διαλόγου, με συμφωνία που ανακοίνωσε και η Κομισιόν και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, μιλάμε επί προεδρίας, ο αρμόδιο ε, προεδρεύοντας τη Δανία, το Συμβούλιο έκανε πίσω. Θα ψηφίσουμε λοιπόν το κείμενο σήμερα ε, όπως συμφωνήθηκε με το Συμβούλιο. Εμεί κάνουμε έκκληση στο Συμβούλιο να τιμήσει το λόγο του. Όπως θα συμφωνήσαμε τέλη Ιουνίου. Εντάξει, του αφήνουμε, να του αφήσουμε κάποιο περιθώριο να συζητήσουμε, αλλά μόνο να συζητήσουμε. Εντάξει, τότε να μην ψηφίσουμε την οριστική το οριστικό κείμενο σήμερα, να μην κάνουμε την τελική ψηφοφορία σήμερα, αλλά δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Ο λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο κάνει πίσω, το κάνει για να μας παρεμποδίσει από το να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τους φορολογικούς παραδείσους, κάτι που είναι έσχος. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λάμπερτς. Ε, θα ψηφίσουμε αυτή την πρόταση πριν ε, περάσουμε στο νομοθετικό ψήφισμα. Θα περάσουμε τώρα στην ε, ψηφοφορία για τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ε, Ο κύριος Σλούτε έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ακούσω τα σχόλια της Κυπριακής Προεδρίας. Τι έχετε σχολιάσει η Κυπριακή Προεδρία από αυτού. Κατανοώ την ερώτηση. Και θα ήθελα να την απαντήσω θετικά, αλλά δεν παριστάτε το Συμβούλιο και ως εκ τούτου δεν μπορεί να απαντηθεί θετικά, καταφατικά η ερώτηση. Έτσι λοιπόν θα πράσουμε στην ψηφοφορία για την ούτως τροποποιηθήσα πρόταση υπέρ. Κατά αποχές γίνεται δεκτή. Τώρα θα ψηφίσουμε για την πρόταση του εισηγητού για αναβολή της οριστικής ψηφοφορίας, τελικής ψηφοφορίας. Υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές γίνεται δεκτή. Καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Λάγκε για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας και του Περού. Υπάρχει μια πληθώρα τροπολογιών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα τις ψηφίσουμε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, τροπολογία 28 με ονομαστική ψηφοφορία, άχελη ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται 32 με, οριστική, με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία υπαριθμών 33 ονομαστική ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται τροπολογία υπαριθμών 34 δέλτα ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα θα έρθουμε στην τροπολογία 35, ονομαστική ψηφοφορία, ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Θα έρθουμε στην ψηφοφορία για την όντως τροποποιηθήσα πρόταση. Περ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Παρακαλώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας για το νομοθετικό ψήφισμα και την αναπομπή στην Επιτροπή για να μπορέσουμε να ε, μπούμε στην συζήτηση του τριμερούς διαλόγου. Λοιπόν, ψηφίσουμε σχετικά με αυτή την πρόταση. Υπέρ παρακαλώ η κατά αποχές εγκρίνεται. Καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση του Γιώργου Λάιχτφριντ για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντρικής Αμερικής οι τροπολογίες του πρώτου μπλοκ εκ μέρους της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Τώρα, στην τροπολογία υπαρχών 37 με ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρθών 31. Ονομαστική ψηφοφορία. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 32. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαρχών 38. Ονομαστική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαρχών 39. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται τροπολογία υπαριθμών 40 δέλτα. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 41. Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τώρα θα περάσουμε στη ψηφοφορία για την ούτως τροποποιηθήσα πρόταση. Πε παρακαλώ. Κατά. Ε, γίνεται δεκτή. Κύριε Σιγητά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ενώπιον της ιδίας κατάστασης όπως ε, στην περίπτωση της Κολομβίας και του Περού. Και θα ήθελα να σας ε, ζητήσω να μην, γίνει, να μην διεξαχθεί η ψηφοφορία μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο και την Επιτροπή και να αναπανθεί στην Επιτροπή μέχρι τότε. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, ψηφίζουμε την πρόταση του συγητού. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλή επιτυχία στις διαπραγματεύσεις σας εύχομαι. Και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Γκέριγκερ Ντεόντενμπουργκ για επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων. Η τροπολογία υπαριθμών 62 της Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έτσι καταπίπτουν οι άλλες τροπολογίες και τώρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία έτσι όπως ε, τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο ονομαστικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία άρχεται ψηφοφορία πέρασε της ψηφοφορίας εγκρίνεται θερμά συγχαρητήρια και τώρα θα περάσουμε στην έκθεση του κυρίου Μορέιρα για τις αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις για το Πακιστάν. Η τροπολογία 47, το κείμενο στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Λοιπόν, η ορθροβηθής πρόταση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα θα περάσουμε στο μαθητικό ψήφισμα με ονομαστική ψηφοφορία, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα ε, για την κατάσταση στη Συρία. Ο κύριος Κονμπεντίτ ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ. Euh, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχω μία προφορική τροπολογία, θα τη διαβάσω αγγλικά για να την καταλάβουν όλοι. Αφορά την παράγραφο 2 και αφορά τους ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Στο κείμενο αναφέρεται θα πρέπει να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσθέσουμε και τις χώρες μέλη έτσι ώστε να υιοθετήσουν μία υπεύθυνη προσθήκη να υιοθετήσουν ανθρωπιστικά μέτρα τους ετούντες άσυλο από την προσθήκη στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ απλή προσθήκη και πιστεύω ότι όλοι οι χριστιανοί, όλοι όσοι πιστεύουν και δεν πιστεύουν θα μπορούσαν να συμφωνήσουν με αυτό. Υπάρχουν ε, στάσεις. Ο κύριος Χαλαφράγκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρα; Θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση σε σχέση με την προφορική τροπολογία που κατέθεσαν οι πράσινοι. Η ομάδα μου συνήθως εκπληρώνει αυστηρά τις ε, δεσμεύσεις που υπογράφει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με τους όρους των διαπραγματεύσεων αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα λάβει τα ενδεδειγμένα και επεύθυνα μέτρα. Και προφανώς μεταξύ αυτών των μέτρων συμπεριλαμβάνονται τα ανθρωπιστικά μέτρα έτσι όπως ανταποκατοπτρίζεται στη συζήτηση που είχαμε με την κυρία Άστον τις προάλλες. Συνεπώς ε, η προσθήκη αυτής της φράσης είναι περιττή και η ομάδα μου αντιτίθεται. Θα πρέπει παρόλα αυτά να πω ότι υπάρχουν 40 βουλευτές που είναι κατά του να γίνει δεκτή αυτή η τροπολογία, άρα είναι επαρκής ε, ο αριθμός. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να γίνει δεκτή η προφορική τροπολογία. Τώρα θα περάσουμε στην τροπολογία παριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία υπαριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Και τώρα θα περάσουμε στο σύνολο του ψηφίσματος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Το ψήφισμα για τη Συρία γίνεται δεκτό. Και τώρα θα περάσουμε στην ψηφοφορία για έξι ψηφίσματα εν σχέση με την χρησιμοποίηση δικαιοσύνη για πολιτικού σκοπού στη Ρωσία. Εδώ δεν έχουν υποβληθεί τροπολογίες. Άρα λοιπόν θα ψηφίσουμε το ψήφισμα στο σύνολό του. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Το ψήφισμα γίνεται δεκτό. Και τώρα θα περάσουμε στην ε, ψηφοφορία για το ψήφισμα της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων για στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση που παρουσιάστηκε χθες. Λοιπόν, θα διεξαχθεί η ψηφοφορία για την αιτιολογική σκέψη Γ. Εδώ έχει ζητηθεί χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Και τώρα θα περάσουμε, περάσουμε θεολογική σκέψη ε, το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. εγκρίνεται και για την αιτιολογική σκέψη έχουμε, πρέπει να ψηφίσουμε σε δύο χωριστά τμήματα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στο δεύτερο τμήμα, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Λοιπόν, το ψήφισμα έτσι όπως έχει τροποποιηθεί. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Υπέ, ε, εποχές, συγγνώμη, δεκτό. Εγκρίνεται. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται εδώ η ψηφοφορία. Και επειδή θα ξεκινήσουμε άμεσα με τις επεξηγήσεις ψήφου, παρακαλώ όσους δεν επιθυμούν να προβούν σε μια επεξήγηση ψήφου να εγκαταλείψουν την αίθουσα το ταχύτερο. Διακόπτεται η συνεδρίαση για